Yeah, yeah. <laughs> Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλώ σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού και σας καλωσορίζω θερμά. Αυτή την εποχή βρισκόμαστε μέσα στη διαδικασία ελέγχου του προϋπολογισμού και πριν ε, μπω στην ουσία θα ήθελα να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Επίτροπο κύριο Σεύκοβιτς, ο οποίος θα απαντήσει και είναι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Επιτροπή μας και τον καλωσορίζουμε. Επίσης ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα ασχοληθούμε με τον τομέα της ειδικότητα του Επιτρόπου που ε, αυτή τη στιγμή έχει συχνότητα λαθών μηδενική. Κανένα λάθος. Οπότε αυτό είναι προς τιμήν μας, διότι πολύ σπάνια μας ε, συγχαίρει κάποιος και συνήθως η κατάσταση δεν είναι τόσο θετική. Δεν τολμώ να πω ότι θα μας συγχαρούν όλα τα μέλη. Μάλλον θα απορρίσουν πώς φτάσαμε και καταλήξαμε σε αυτή ε, την, το μηδενικό ποσοστό σφαλμάτων. Αλλά ακόμα και αν υπάρχουν σφάλματα είναι πάρα πολύ χαμηλά, πολύ λίγα. Και ως Επιτροπή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να διευθετήσουμε το θέμα σωστά και με την Κομισιόν έτσι ώστε να προσανατολιστούμε από ένα προϋπολογισμό περιεχομένου σε ένα προϋπολογισμό εκτελεστικό και έχουμε ήδη μελετήσει από την Κομισιόν ε, τις για τη διαχείριση του προϋπολογισμού και τις εκθέσεις του κ. Μούλντε, το θέμα της λογοδοσίας και της περαιτέρω συμμετοχής και συμβολή των κρατών μελών. Χαιρετίζω επίσης και τους εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καλωσορίζω τον κύριο Τομέ Μουγκουρούζα, σε αυτό το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αλλά προηγουμένως ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν τίποτα επισημίες για να τροποποιήσουμε τη ημερήσια διάταξη. Όχι λοιπόν, δεν υπάρχουν. Ε, έχει λοιπόν αρχίσει τώρα επισήμως η συνεδρίαση, έχουμε τις ε, διερμηνίες που χρειάζονται και επίσης μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Και ε, έρχομαι κατευθείαν στο σημείο 3, το πρώτο προσυζήτηση ε, και θα ήθελα πριν δώσω το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο, θα ήθελα να καλωσορίσω και μία ομάδα επισκεπτών από την ε, πόλη μου και είναι μέλη, νέα μέλη, η νεολαία της ομάδας του πολιτικού κόμματος των φιλελευθέρων της περιφερειάς μου. Και δίνω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου, κύριο Τομέ Μουγκουρούζα. Α, δεν κλείνει. Δεν κλείνει. Members of the Budgetary Control Committee, dear Commissioner, chapter... Το κεφάλαιο 9 παρουσιάζεται η αξιολόγηση των δαπανών αυτού του θεσμικού οργάνου και άλλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα πολιτικής αντιπροσωπεύει 7% των δαπανών που έγιναν το 2011 δαπάνες για ανθρώπινους σπόρους όπως είναι οι αποδοχές, ε, ε, δαπάνες για κτίρια, ενέργεια, επικοινωνίες και τεχνολογική πληροφορική. Για το σκοπό του ελέγχου το 2011 το ελεγκτικό συνέδριο εισήγαγε τρεις ε, βασικές βελτιώσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτα την βελτίωση που σχετίζεται με τον αριθμό των συναλλαγών των ελεγκτών που καλύπτουν τις ε, δαπάνες των θεσμικών οργάνων. Το 2011 το δείγμα το οποίο ελέγχθηκε από το συνέδριο ήταν 151 συναλλαγές, ενώ το 2012 ελέγχθηκαν 56 συναλλαγές. Η δεύτερη βελτίωση αφορά την εναρμόνιση της προσέγγισης όσον αφορά τα σφάλματα προμηθειών και τα αντίστοιχα κεφάλαια στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Από το 2012 υπήρξαν σοβαρά σφάλματα στη διαδικασία αυτή, τα οποία διαπιστώθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο. Η τρίτη βελτίωση, η οποία εισήχθη από το συνέδριο το 2012, αναφέρεται στον έλεγχο των εποπτικών συστημάτων των των, των θεσμικών, του ελέγχου των θεσμικών οργάνων. Και εδώ το ελεκτικό συνέδριο κάνει μια εισβάθος εξέταση δύο θεσμικών οργάνων αναέτος ε, ε, εκ περιτροπής και η εξέταση καλύπτει τους ανθρώπινους πόρους και τις διαδικασίες ε, προμηθειών. Το 2012 ο έλεγχος των θεσμικών οργάνων αφορά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η έκβαση είναι, το αποτέλεσμα είναι θετικό και το συνέδριο καταλήγει ότι οι συναλλαγές και οι δαπάνες, οι διοικητικές δαπάνες το 2012 ε, ήταν ε, κανονικές. Το συνέδριο βρήκε ότι μόνο από μία από τις 151 συναλλαγές που ελέγχθηκαν είχε επηρεαστεί από κάποιο σφάλμα και κατά πάσα πιθανότητα ε, και το ποσοστό αυτό των σφαλμάτων είναι περίπου 0%. Επίσης καταλήγει ότι ε, το Απτικό Συμβούλιο ακολουθεί τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού ε, του, του κανονισμού. Το συνέδριο εξέτασε εις βάθος τα εποπτικά συστήματα. Ωστόσο υπάρχουν κάποια μικρά σφάλματα σε κάποιες διαδικασίες προμηθειών και στην ε, διαχείριση των ε, κοινωνικών επιδομάτων. Στη βάση των συμπερασμάτων το συνέδριο συνιστά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι οι αρχές ε, να εξασφαλίσουν την συμβατότητα των διαδικασιών ε, προμηθειών. Αγαπητά μέλη, εγώ βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση που έχετε και σε ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Τομέ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μάρκους Πίπερ, εισηγητή του θέματος. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να συζητήσουμε την εσωτερική διοίκηση ενδελεχώς και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι βάσει των δεδομένων του ελεγκτικού συνεδρίο από το 0,1% των σφαλμάτων πήγαμε στο 0,0%. Όμως θα ήθελα να θέσω και ορισμένα ερωτήματα τα οποία ήδη έχουν τεθεί και από ορισμένους συναδέλφους. Πρόκειται ιδιαίτερα για τη μη τήρηση της διαδικασίας για τους δημόσιους διαγωνισμούς, δημόσιες προμήθειες, επίσης για την επιλογή υποψηφίων για υπαλλήλων, για τους μισθούς, ύψος των μισθών και για μας είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιες είναι οι διατάξεις ε, για τους ε, υπαλλήλους, για την κατάρτισή τους και τα υπάρχοντα προβλήματα και την υπόθεση Τσίγκλερ. Καταρχάς, λοιπόν, για ε, την τελευταία απαλλαγή το πρώτο θέμα λοιπόν, οι διατάξεις για το προσωπικό, για τους υπαλλήλου. Εδώ στην τελευταία απόφαση του Κοινοβουλίου είπαμε, στο τελευταίο ψήφισμα είπαμε ότι έχουμε ορισμένες ερωτήσεις όσον αφορά το μισθολόγιο, τον πίνακα μισθολογίου, τις ε, ε, προσωρινές ε, συμβάσεις και τις έκτακτες συμβάσεις. Μας έδωσαν λοιπόν ορισμένες απαντήσεις, αλλά αυτό που ακόμα δεν, δεν έχει απαντηθεί είναι ότι υπάρχουν σαφείς δομές, αλλά στην κινητικότητα των υπαλλήλων, ιδίως των υψηλότερων στελεχών, η Κομισιόν έχει ένα ευρύτατο περιθώριο εσωτερικής ε, ε, διακριτικής ευχέρειας. Ε, ποιον προτιμάει, πώς θα ταξιδέψει, ποιος θα ταξιδέψει, που θα μείνει και τέτοιες λεπτομέρειες. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε ποια κριτήρια τηρούνται και αν υπάρχουν σαφείς διατάξεις για τα υψηλότερα στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη ή αν υπάρχει ένα ευρύ περιθώριο ευελιξίας. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την κατάρτιση των υπαλλήλων Εμένω λοιπόν ε, στο θέμα του προσωπικού των υπαλλήλων. Έχουμε ένα πρόγραμμα εξέλιξης ε, των υπαλλήλων το οποίο είναι πολύ δαπανηρό. Ε, βεβαίως στοχεύουμε στην ποιότητα. Η Ευρώπη στοχεύει σε ποιοτικού υπαλλήλους, σε ποιοτικά στελέχη. Όμως, όσον αφορά το, τη σχέση κόστους-οφέλους αυτών των προγραμμάτων εξέλιξης, έχουμε το εξής ερώτημα έχει αντιπαραταθεί αυτό με μια άλλη παρόμοια δομή. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνετε εσείς ως κατάρτιση και ποια σχέση κόστους ωφέλους υπάρχει μεταξύ του κόστους κατάρτισης και των ωφελών των υπαλλήλων. Εν συνεχεία... Stehen, nicht Διαδικασίες πρόσληψης ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι γίνεται με τους συμβασιούχους και πώς τους προσλαμβάνεται βάσει πριν ποιοτικών κριτηρίων και ε, έχω μία ερώτηση εδώ, ένα, ένα ζήτημα και ε, προς το ελεγκτικό συνέδριο. Ο διαγωνισμός, οποίος, τον οποίο πρέπει να περάσουν όταν ε, θέλει κανείς να γίνει υπάλληλο ή ανώτερο στέλεχος, πιο υψηλό βαθμό. Είναι ένας διαγωνισμός τον οποίο οργανώνει η Κομισιόν. Είναι ο ίδιος ε, διαγωνισμός που πρέπει να περάσουν όταν θέλουν να γίνουν διοικητικοί υπάλληλοι υπάλληλοι στο ελεγκτικό συνέδριο. Έχει δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο μία ξεχωριστή διαδικασία διαγωνισμών για την πρόσληψη υπαλλήλων υπάρχουν διαφορές ή το, η Κομισιόν και το Ελεγκτικό Συνέδριο παίρνει το προσωπικό που χρειάζεται από την ίδια δεξαμενή βάση του ιδίου διαγωνισμού. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση αυτή. Και τέλος υπάρχουν ορισμένε ερωτήσεις που έχουν τεθεί από συναδέλφους. Ο κύριος Τόιρερ από το 19 Απριλίου σε μια επιστολή του 19 Απριλίου 2013 τόνισε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι συγκρούσει συμφερόντων και είπατε, απαντήσατε ότι η, ο Μισελ Πετή που ονομάστηκε ξανά μέλος της Επιτροπής Ad Hoc δεν αντιπροσωπεύει μία σύγκρουση συμφερόντων και η Επιτροπή αυτή Ad Hoc θα πρέπει να εξετάσει την συνεργασία με προηγουμένων επιτρόπων σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ποιες είναι οι προϋποθέσεις με τις, τις οποίες έθεσε η Κομισιόν στον κύριο Μισελ Πετή και ε, κατά πόσον εσείς συμβάλλατε στην αποφυγή μια σύγκρουση συμφερόντων με την επιλογή του. Δεύτερον, γιατί η Κομισιόν αποφάσισε να επιμικίνει, ε, να, παρατείνει τη σύμβαση του κυρίου Μισελ Πετή, ενώ εσείς στην επιστολή σας είπατε και παραθέτω πάλι ότι εδώ και ε, ε, πρόσφατα υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις όσον αφορά τη συμπεριφορά του κυρίου Πετή στην υπόθεση Ντάλι. Ε, ρωτώ λοιπόν για την επιτροπή αυτή, για την επιτροπή έτη, ad hoc δηλαδή δεν υπήρχαν άλλοι υποψήφοι, ήταν ο μόνος, ήταν ο μοναδικός και αν ήταν, ε, υπήρχαν άλλοι βάσει ποιων κριτηρίων αποφάσισαν την επιλογή του Μισελ Πετή. Εν συνεχεία στο ερώτημα 21 που έχουμε θέσει προς τον κύριο Πίμπαλς, Πρόκειται και πάλι για σύγκρουση συμφερόντων και η Κομισιόν απάντησε ότι έχει μόνο χρησιμοποιήσει από την IMG έναν ιδιωτικό σύμβουλο ο οποίος έλαβε ειδική άδεια για τις δραστηριότητε της, για την εργασία του βάσει του άρθρου 16 συνάδει δηλαδή με το άρθρο 16 με την προϋπόθεση ότι δεν θα πρέπει να λάβει άλλες επιδοτήσεις ή περαιτέρω συμβάσεις στα πλαίσια αναθέσεων της Γενικής Διευθύνσεως ΔΕΦΚΟ. Αυτή ήταν η απάντηση κυρίου Πίμπαλς και οι χώρες της ε, Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής, ε, Παλαιστίνη, Μολδαβία, την Ισία, Ουκρανία, ε, αυτές οι χώρες καλύπτονταν από την, την, πρόσληψη αυτού του συμβούλου από την IMG και ήθελα να πω, να ρωτήσω γιατί αναφέρονται ειδικά όλες αυτές οι χώρες στη σύμβαση γιατί και με ποιες προδιαγραφές επιλέχθηκε και γιατί η IMG ως εταιρεία International Management Group χρησιμοποιείται και πάλι ως εμπειρογνώμονες στο θέμα της ε, προστασίας του περιβάλλοντος, του κλίματος. Και 5,5 εκατομμύρια ευρώ έλαβε το 2012. 1,5 εκατομμύριο ευρώ για ένα πρόγραμμα στην, στο Μιανμάρ ενώ ο πρώην υπάλληλος κομισιόν που είχε το φάκελο στα χέρια του α, δουλεύει από το 2011 στη Γενική Διεύθυνση κλίμα, ε, Περιβάλλοντος, Κλίματος. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω γιατί αναφέρονται όλες οι άλλες χώρες σε αυτό το μακρύ κατάλογο χωρών στην απάντηση του κυρίου Πίμπαλς. Λοιπόν, ε, με την μηδενική αυτή, το μηδενικό ποσοστό σφαλμάτων ε, καταλαβαίνετε ότι εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι στο Κοινοβούλιο και αναμένουμε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ ε, για τα εισαγωγικά σας λόγια και θα ήθελα να παρακαλέσω εσάς κύριε πίτροπε να λάβετε θέση από τη δική σας κοπιά και στη συνέχεια θα θέλαμε να αρχίσουμε τη συζήτηση με τους συντονιστές. Κύριε Επίτροπε έχετε το λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αναφέρομαι και στους νέους από τη Βάδη Νιρεμέργη που βρίσκονται εδώ πέρα αυτή τη στιγμή και που είναι πολύ σημαντικό το ότι μπορούν και ενδιαφέρονται για τα ζητήματα ελέγχου της χρησιμοποίηση των κοινοτικών δαπανών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται αυτός ο χρηματοοικονομικός έλεγχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσετε για τη συζήτηση αυτή για την απαλλαγή 2012. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τόμε Μουγκρούζα για την πρώτερη παρέμβασή του και γενικότερα να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να έχουμε ένα τόσο χαμηλό ποσοστό σφάλματο. Αυτό έχει να κάνει με τι πολύ συστηματικέ ανταλλαγέ απόψεων και πυρογνωμοσύνη που έχουμε με το ελεγκτικό συνέδριο και του ελεγκτέ του. Διαδικασία που βοηθάει πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει ένα ύψιστο επίπεδο διοικητική διαχείριση και από πολιτική όμω πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και αυτό ο ανεξάρτητο αυτόνομο έλεγχο που γίνεται από το ελεγκτικό Συνέδριο. Να ευχαριστήσω όμω, Πρόεδρε, και τη δική σα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή όλος ιδιαιτέρως γιατί ε, εν προκειμένου εκπροσωπείτε εσείς το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παραγωγική σας, ε, τον παραγωγικό σας έλεγχο, την πίεση που ασκείτε, την επικοδομητική συνεργασία την οποία έχουμε μαζί σας που είναι πάρα πολύ σημαντική είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να απαντούμε στις πολύ εύστοχες ερωτήσεις που τίθενται από τη δική σας την Επιτροπή και προσπαθήσαμε, όπως είδατε, να απαντήσουμε στις 50 περίπου ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή σας όσον αφορά τη δικασία απαλλαγής 2012. Θα ήθελα προφανώ να απαντήσω στα επιμέρου ερωτήματα που έθεσε ο εισηγητή, αλλά θα ήθελα να αφαιρθώ πρώτα σε δύο σημαντικά ζητήματα. Προετοιμαζόμενο για τη συνεδρίαση αυτή, μου προτάθηκε να αναφερθώ στα δύο αυτά ζητήματα όσον αφορά την εισαγωγική μου παρέμβαση. Όσον αφορά καταρχάς την, παρέμβαση, την μεταρρύθμιση με συγχωρείτε του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καταφέραμε πολύ γρήγορο να ολοκληρώσουμε τις πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και χάρη στην νέα αυτή συμφωνία πολλά πλέον πράγματα γίνονται πολύ πιο σαφή όπως και η εξοικονόμηση η οποία απορρέει από τη μεταρρύθμιση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ όσον αφορά το διοικητικό προπολογισμό από σήμερα μέχρι το 2020 και 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή η μεταρρύθμιση, κυρίω η μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού προγράμματος αρχίσει να λειτουργεί πλήρω. Πώς καταφέραμε να πετύχουμε τη σημαντικότατη αυτή εξοικονόμηση, καταρχάς μείωση 5% όσον αφορά το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταρρύθμιση που θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Να πω επίση ότι Πέρασαν 9 χρόνια από τότε που κάναμε τι άλλε σημαντικέ μεταρρυθμίσει όσον αφορά τον κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που είχαμε μια πολύ θετική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καταφέραμε κατά αυτόν τον τρόπο να επιφέρουμε νέε σημαντικέ διαρθρωτικέ ε, αλλαγέ στον κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση, ιδίω όσον αφορά το συνταξιδοτικό σύστημα, μολονότι το όλο εγχείρημα ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκο, καταφέραμε πιστεύω αρκετά αρμονικά να πετύχουμε τη μεταρρύθμιση αυτή χωρίς σε καμία περίπτωση να ταραχθεί η λειτουργία του όλου συστήματος. Ξέρετε επίση ότι για δύο χρόνια, 2013-2014, έχουν παγώσει οι συντάξεις και οι μισθοί επίσης περνάμε σε μια εργάσιμη εβδομάδα 40 ωρών, μία από τις πιο εντατικά εργασιακές εβδομάδες όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, καταφέραμε όμω να διατηρήσουμε τα βασικά στοιχεία τα οποία εξασφαλίζουν την ύψιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από του υπαλλήλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά ανταποκρίνονται στο πολύ σημαντικό θεματολόγιο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θα έχουμε μία μείωση 5%, δηλαδή 1% τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι το 2017 όσον αφορά το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πράξη τι σημαίνει αυτό, ότι 250 θέσεις εργασίας ήδη από του χρόνου θα καταργηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το θεσμικό όργανο που προβλέπει τις λιγότερες νέες θέσεις εργασίας για τα επόμενα χρόνια. Ακούσαμε τις δικές σας συμβουλές και είχαμε και συζητήσει με την κυρία Κρέσλερ για να καταφέρουμε να βελτιώσουμε το σύστημα ελέγχου που έχουμε, πώς μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα ετήσιου ελέγχου όσον αφορά το έργο των επιτρόπων, πώς μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα όλο το υποστηρωτικό προσωπικό που πλαισιώνει τους επιτρόπους, καθώς επίσης και όλους τους εμπειρογνώμονες και δήμονες που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα, θα έρθω και στο σημείο αυτό, ξέρω ότι ανήκει σε ερωτήσεις σας και το σημείο αυτό. Εξίσου επίσης σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι αυτή η διαδικασία ελέγχου και επιτήρησης ε, καταδεικνύει τελικά το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βοηθήσει και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, γιατί παρέχουμε προς τα άλλα θεσμικά όργανα πολύ σημαντικές υπηρεσίες. Και ουσιαστικά αυτό αντιστοιχεί επί του παρόντος σε 1.700 θέσεις ισοδύναμης πλήρης απασχόλησης. Κατά αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να κάνουμε πολύ σημαντική εξοικονόμηση για τον κοινοτικό προπολογισμό και βέβαια βλέπουμε ότι ένα 22,5% των συνολικών θέσεων εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013 είχαν να κάνουν με υπηρεσίες ε, υποστήριξης. Και όταν μιλούσαμε με την κυρία Κρέστλερ το ποσοστό αυτό ήταν 30%. Βλέπετε ότι έχουμε καταφέρει να το μειώσουμε. Θα καταφέρω να σας δώσω όμως και πιο συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία λίγο αργότερα στην παρουσίασή μου. Τώρα, πώς θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε σε νέες προτεραιότητες και νέους στόχους. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και άλλα θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε φορά που προκύπτουν νέες αρμοδιότητες, συζητάω πάντα με τους συνεργαζόμενούς μου για να δούμε τελικά πώς θα καταφέρουμε να καλύψουμε τις νέες αυτές αρμοδιότητες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι από το να προσλαμβάνουμε νέους ανθρώπους να κατανέμουμε καλύτερα, να κάνουμε έναν καλύτερο επιμερισμό του υφιστάμενου προσωπικού. Η αρχή αυτή θα εμπνέει την πολιτική μας για το προσωπικό τα υπόλοιπα χρόνια και πιστεύω ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Πρέπει να διοργανώσουμε όμως πολλές υπηρεσίες μας. Ήδη δημιουργούμε υπηρεσίες υποστήριξης κοινέ για πολλές γενικές διευθύνσεις, παρέχουμε υπηρεσίες κοινέ και προς άλλα θεσμικά όργανα, προσπαθούμε να έχουμε καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες διαδικασίες όσον αφορά την πληροφορική, και κατά αυτόν τον τρόπο κάνουμε εξοικονόμηση τόσο σε χρηματοοικονομικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό. Να κάνω τώρα και κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τις αποκεντρωμένες αυτές υπηρεσίες και οργανισμούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την κυρία Γκρέσλερ και με άλλα μέλη της Επιτροπής μας, της Επιτροπής σας, με συγχωρείτε, εδώ και πάρα πολλή χρόνια ασχολούμεθα με το ζήτημα αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι η εργασία που επιτελέσαμε ήταν σημαντικότητη. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι ε, αυξήθηκε σημαντικότατα ο αριθμός των αποκεντρωμένων αυτών οργανισμών. Ο πρώτος δημιουργήθηκε το 1975, 10 το 2000 και έχουμε φτάσει σε 30 τέτοιες υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά περίπτωση έγινε η ανάπτυξη των οργανισμών αυτών με βάση τις ανάγκες μας δηλαδή και επομένως ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα καταφέρουμε να διαχειριστούμε με έναν ενιαίο και κεντρικό τρόπο τις νέες αυτές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βλέπω ότι έχουμε πλέον μια κοινή προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις αποκεντρωμένες αυτές υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποτελέσει η νέα αυτή προσέγγιση ένα σημείο αναφοράς προκειμένου να οργανώνονται ενιαία εναρμονισμένα όλα τα επόμενα χρόνια οι νέες υπηρεσίες οι οποίες θα δημιουργηθούν. Επ' αυτού όμως χρειάζομαι και τη δική σας την υποστήριξη, τη δική σας τη συμβολή, τη δική σας την πολιτική καθοδήγηση. Γιατί γνωρίζω ότι ένας από τους σαφείς στόχους της κοινή αυτής προσέγγισης ήταν να δούμε κάθε φορά ποιες είναι οι δυνατότητες συγχώνευσης συνεργειών προκειμένου να καταφέρουμε να καταστήσουμε το έργο των υπηρεσιών αυτών όλο και πιο διαφανές. Και όντως έγινε μια τέτοια συγχώνευση. Η ΣΥΠΟΛ και η Europol και οι δύο αυτές υπηρεσίες όπως το ξέρετε ασχολούνται με το ίδιο πεδίο αρμοδιότητας, δεν έχουν ακριβώς την ίδια ατζέντα, πάντως ε, ε, έχουν να κάνουν με την αστυνομική κατάρτιση και την αστυνομική συνεργασία. Κάναμε λοιπόν κάποιους πολύ σημαντικούς ακριβείς υπολογισμούς και συνειδητοποιήσαμε ότι αν συγχωνεύαμε τις δύο αυτές υπηρεσίες θα καταφέρναμε να πετυχαίναμε έναν πολύ σημαντικό εξορθολογισμό του προσωπικού και μια πολύ σημαντική εξοικονόμηση όσον αφορά τον προπολογισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή σας η οποία στήριξε την προσέγγιση αυτή. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί γιατί δυστυχώς ε, η πρόταση αυτή δεν είχε την περαιτέρω υποστήριξη τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολό του όσο και την υποστήριξη του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ε, δεν τα βάζει κάτω. Θα συνεχίσουμε αυτή την διοργανική προσέγγιση και θα προωθήσουμε περισσότερο και άλλες διοργανικές συμφωνίες θα δημιουργηθεί επίσης και μια διοργανική ομάδα η οποία θα έχει ως στόχο να καταφέρει να ανακαλύψει και άλλες περιπτώσεις ε, όπου θα μπορούσαμε να συγχωνεύσουμε υπηρεσίες ή να πετύχουμε συνέργειες. Η συμφωνία πάντως αυτή που ήδη επετεύχθη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς που θα, διέπει, που θα χαρακτηρίζει πλέον τον τρόπο με τον οποίο θα εργάζονται και θα δημιουργούνται στο μέλλον οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να είναι όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικές. Τέλος, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αρχίζω και απαντώ σιγά σιγά και στις ε, ερωτήσεις που έθεσε ο εισηγητής σας το ζήτημα της ε, πρόληψης και της διαχείρισης ε, της σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρω ότι τα ερωτήματά σας είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο δημοσιονομικός κανονισμός και ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπουν πολύ σημαντικά μέτρα για το μετριασμό των συγκρούσεων συμφερόντων και πιστεύω ότι έχουμε πετύχει πολύ σημαντικές βελτιώσεις στο μεταρρυθμισμένο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Θα έχουμε όμως και κατευθυντήρες γραμμές σύντομα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καλύψουμε και το προσωπικό και τους υπόλοιπους φορείς που εργάζονται στα πλαίσια των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιοι είναι τα νέα αυτά μέλη. Είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διοικητικών Συμβουλίων που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις που προβλέπονται αυτή τη στιγμή, μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών καθώ καθώς επίσης και άλλα μέλη των ε, Συμβουλίων Προσφυγής. Έφεσης. Κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε όλο το προσωπικό, όλα τα μέλη, όλους τους συνεργάτες των ε, υπηρεσιών, των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούν όλοι τους ενιαίους, ενιαίους αυτούς κανόνες που διέπουν την, ε, το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων. Θα σας στείλουμε λοιπόν πολύ σύντομα τους εναρμονισμένους αυτούς κανόνες και τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές και ξέρω ότι η Επιτροπή σας προβλέπει ήδη από τον Ιανουάριο 2014 μία έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσετε κι εσείς να συμβάλλετε πάρα πολύ στην όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου να καταφέρουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το εφιστάμενο σύστημα. Ολοκληρώνοντας την αρχική μου αυτή παρέμβαση, θα ήθελα να πω ότι ελπίζω ότι καταφέραμε να σας πείσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε δεδομένο το γεγονός ότι θα έχουμε μια καλώς λειτουργούσα διοίκηση και διαφανή διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταυτού προσπαθούμε κάθε φορά να καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια, να βελτιωθεί η ιδεοντολογία, και μέσω της εργασίας μας αυτής θέλουμε να καταδείξουμε επίσης ότι θέλουμε σε κάθε περίπτωση να αποτελεί η κοινοτική διοίκηση θέμενη αξία για τον Ευρωπαίο πολίτη και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποια από τα ερωτήματα τα οποία έθεσε ο Αλλά παρακαλώ θυμίστε μου αν ξεχάσω κάτι. Όπως Τη σημείωσα τις ερωτήσεις λοιπόν. Έχουμε το θέμα έψο που είναι ο φορέας, το Ίδρυμα, το διαθεσμικό, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο την Κομισιόν, παρόλο εμείς είμαστε οι βασικοί πελάτες, αλλά και άλλα ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι λοιπόν ε, ένας φορέας που εξυπηρετεί όλα τα θεσμικά όργανα. Εάν τώρα αλλάξουμε το σύστημα προσλήψεων, ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε δίκαιοι και ότι προσλαμβάνουμε τους βέλτιστους για τις θέσεις που χρειαζόμαστε με τις ε, ε, σωστές προδιαγραφές και με τη σωστή περιγραφή των δεξιοτήτων που απαιτούνται για κάθε εργασία. Έχουμε τώρα εισαγάγει αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης που αποδίδει πολύ καλύτερα από μια συνέντευξη μισής ώρας διότι έχουν όλες τις δυνατότητες να αξιολογήσουν τα κριτήρια, παραδείγματος χάρη ε, την εργασία μέσα στο όλο εργασιακό περιβάλλον, ε, τα προσόντα του κλπ. και να κρίνει ότι αυτός είναι ο καλύτερος υποψήφιος, ο καλύτερος υπάλληλος. Επίσης έχουμε τους, τους ε, διαγωνισμούς αυτούς, τα τεστ αυτά που κάνουμε βάσει του, της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά τα τεστ αυτά Συνήθω γίνονται για γενικό προσωπικό την άνοιξη, το υποστηρικτικό προσωπικό το καλοκαίρι και μεταφραστές το φθινόπωρο. Ε, όσον αφορά τη συγκεκριμένη σας ερώτηση για το πώς προσλαμβάνουμε ειδικού, παραδείγματο χάρη ε, ελεγκτικό προσωπικό. Κάνουμε συγκεκριμένες, συγκεκριμένους διαγωνισμούς για τους ελεγκτικούς φορείς, διότι όπως ξέρετε δεν είναι μόνο το ελεγκτικό συνέδριο που χρειάζεται ελεγκτές, αλλά ε, όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παρόμοιες ανάγκες και κάθε γενική διεύθυνση. Όσον αφορά τις αποστολές, εδώ είναι σαφές ότι υπάρχουν οδηγίες στον κανονισμό περί αποστολών, οι κανόνες εφαρμόζονται ισότιμα σε όλους, το ίδιο, η ίδια οροφή για τα ξενοδοχεία και ορισμένες παρακλήσεις είναι δυνατόν να γίνουν, αλλά είναι σπάνιες όταν αναφέρομαι σε παρεκκλήσεις, σε παραδείγματος χάρη, όταν πρέπει Κάποιο να βρίσκεται σε κάποιο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή να διαμείνει, η οποία είναι ασφαλής ε, όταν υπησέρχονται θέματα ασφάλειας δηλαδή και δεν μπορεί, δεν έχει άλλες επιλογές. Πρέπει όμως η παρέκκληση να δικαιολογείται ε, και να είναι ευλογή. Τώρα, για ε, το μέλλον είναι πολύ σημαντικό πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε όχι μόνο τον έλεγχο των κονδυλίων αν έχουν οι πιστώσεις αυτές ε, ε, δαπανηθεί σωστά αλλά και όλη τη διαδικασία Παραδείγματο χάρη ένα αεροδρόμιο έχει χτιστεί ε, με δημόσιο διαγωνισμό. Εφαρμόζονται οι δημοσιονομικές και κανονισμοί του προϋπολογισμού. Εντάξει, αλλά πρέπει επίσης να κρίνουμε τελικά το όφελος, αν ήταν μια καλή επένδυση. Ε, οπότε αυτά τα στοιχεία απαιτούν μια πολύ πιο περίπλοκη αξιολόγηση. Έχουν πολύ περισσότερες ε, πτυχές αξιολόγησης. Πιστεύω ότι αυτά θα εφαρμοστούν στο μέλλον για τα κεφάλαια 1 έως και 4. Για το κεφάλαιο 5 και απαντώντας στον εισηγητή σας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα κριτήρια για την απόδοση ε, ενός υπαλλήλου θα πρέπει να ε, βασιστούν, να, να, κρίνουν και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης του υπαλλήλου. Όταν ήλεγχα τις δαπάνες για την κατάρτιση, την εκπαίδευση και το πώς, ε, τι, τι δαπανούμε για ποια κατάρτιση και πώς σα στελέχη εκπαιδεύτηκαν κλπ, πώς οι υπάλληλοι, δεν θα εκπλαγείτε ότι οι περισσότερες μέρες κατάρτισης, 8 με 11 ε, τις είχαμε διαθέσει για κατάρτιση ελεγκτών, διότι υπάρχει ένας νέος δημοσιονομικός κανονισμός και χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση ε, των ελεγκτών και πιστεύω το αποτέλεσμα του ότι έχουμε εξαιρετικά έμπειρους ελεγκτές δικαιολογεί την κατάρτιση και προσφέρει προστιθέμενη αξία ε, για τα χρήματα που δαπανούμε. Σχετικά τώρα με το, τη σύγκρουση συμφερόντων θα είμαι πολύ ειλικρινής για, το, το ζήτημα της επιστολής του κυρίου Πίμπαλς ε, και όσον αφορά αυτή την εταιρεία, την IMG, δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Ε, δεν μπορώ να σας πω κασίες, ή ε, στοιχεία από το κεφάλι μου χωρίς να έχω μια βάση δεδομένων. Ε, σας διαβεβαιώνω όμως ε, ότι ε, εάν υπάρχει σαφής λόγος να εξετάσουμε το θέμα αυτό περισσότερο σε βάθος, θα το κάνουμε είτε μέσω της διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, είτε με κάποια άλλη ειδική διεύθυνση. Τώρα, για την επαναπρόσληψη του κυρίου Πετή, αυτό συζητήθηκε και από τον Ευρωπαίο μεσολαβητή με μένα. Ε, γνωρίζω σαφώς ότι η Επιτροπή Διοντολογίας θα εξετάσει πολλές περιπτώσεις ανανέωσης θητείας ε, και ε, νέες υποψηφιότητες, ε, ορισμένοι επίτροποι θα φύγουν, άλλοι θα έρθουν, άλλοι θα ολοκληρώσουν την εργασία τους για την Κομισιόν. Οπότε αντιλαμβάνουμε σαφώς πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα της απόδοσης και των εργασιών αυτή τη Επιτροπή Δεοντολογία. Θα είναι λίγα σημαντική του χρόνου. Και σα διαβεβαιώ ότι όλα αυτά τα έχω σημειώσει και θα τα συζητήσω στην έδρα μου, στην Κομισιόν και θα δω με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε όταν φτάσει η κρίσιμη αυτή η περίοδος όπου θα χρειαστεί η παρέμβαση ε, της Επιτροπής Δεοντολογίας η απόδοση της και το όλο έργο της θα εκτελεστεί με τον βέλτιστο τρόπο έτσι ώστε να μην δημιουργήσει καμία ε, ανησυχία ή επιφύλαξη ως προς το έργο της. Εν συναχεία, συγγνώμη πρόεδρε, έχω διάφορες σημειώσεις από εδώ και από εκεί. Απρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συντονιστές των ομάδων. Και να αρχίσουμε με την κυρία Γκρέσλερ από το ΕΡΚ. Α, συγγνώμη. Θα, επανέλθω, λέει ο θα σα δώσω στοιχεία συγκεκριμένα. Ναι, είναι μια μακρά διαμάχη σε σχέση με αυτούς τους αριθμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προθυμία που δείξατε να έρθετε πάλι εδώ και σε ευχαριστούμε επίση πολύ για τι ε, απαντήσεις σας που τελικά δεν τι ε, δεν τις ερμηνεύσατε κακόπιστα. Αντιθέτως, όσον αφορά τον κύριο, ε, όσον αφορά τον κύριο Πιτ, σε μία επιστολή στις 11 Ιουλίου του 2013 μας είπατε ότι ο κύριος Πετή δεν είχε κανέναν ρόλο σε όλη αυτή την την υπόθεση του Επιτρόπου Ντάλι. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Σε 8 και 9 Μαΐου έγινε μια τηλεφωνική επαφή με τον κύριο Πετή όσον αφορά την διαχείριση αυτής της ε, περίπτωσης. Άρα αυτό δεν ευσταθεί. Θα ήθελα να μου αναφέρετε το δικό σας ρόλο στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής, όταν λέτε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως παρεμβολή μεταξύ της Επιτροπής Δεοντολογίας και αυτού που κάνει σήμερα ο κύριος Πετή, δεν ισχύει. Ε, περίπου 20 επίτροποι θα εγκαταλείψουν την Επιτροπή. Ε, και, και ίσως ε, εσείς ε, θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να περάσετε πάλι μέσα από, ε, την ακρόαση του Κοινοβουλίου και θα φτεθεί το ζήτημα του κυρίου Πετή. Το ερώτημα είναι γιατί λοιπόν διορίστηκε πάλι ο κύριος Πετή όπου υπάρχει μια εξόφθαλμη σύγκρουση συμφερόντων. Εδώ υπό την τωρινή του ιδιότητα ε, στην Επιτροπή σε σχέση με, τις, με τη διατησία ή τις συμφωνίες για τον καπνό. Άρα λοιπόν χρησιμοποιεί το κύριος ε, Πετή για να αποφανθεί για θέματα που αφορούν τον παλαιό του εργοδότη. Άρα λοιπόν, εάν αυτό είναι το μοντέλο που θα ισχύσει για τους μελλοντικούς επιτρόπους, ε, και για την αξιοποίησή τους νομίζω ότι θα υπάρξουν μεγάλες αντιρρήσεις εκ μέρους του Κοινοβουλίου σε σχέση με την, ε, με την Επιτροπή και την μελλοντική της σύσταση. Λοιπόν, θα ήθελα να μας απαντήσετε γιατί ε, διορίστηκε και πάλι ο κύριος Πετή, γιατί πριν από τα Χριστούγεννα του 2012 υπήρξε η δυνατότητα να καταργηθεί αυτή η πραγματικά προβληματική δομή, αν θέλετε, εντός του, της Τώρα, ε, ο, κανονισμός, η υπερσιακή κατάσταση ε, δίνει λαβή σε πάρα πολλές ε, διαμάχες. Ε, μάθαμε ότι η Κομισιόν ασφάλισε δύο Βέλγους υπαλλήλους βάσει του βελγικού ασφαλιστικού δικαίου. Οι στατιστικές που μας στείλατε εσείς τώρα και τις χρησιμοποιεί η Γενική Διεύθυνση ή όχι γιατί βλέπω ότι όσον αφορά τους εκτελεστικούς φορείς, εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί υπάλληλοι οι οποίοι προέρχονται από αυτή την εταιρεία. Τώρα, όσον αφορά την αξιολόγηση όλου αυτού του μοντέλου λειτουργίας, δηλαδή να προσλαμβάνονται στο δημόσιο κάποιοι εργαζόμενοι από τρίτες εταιρείες, ε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι θεμητό να προσφεύγει η Κομισιόν σε τέτοιου είδους ε, μηχανισμούς. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια, πρόκειται να αλλάξετε αυτή την κατάσταση ε, με αυτούς τους προσωρινά εργαζόμενους, του οποίους προσλαμβάνετε από άλλες εταιρείες. Τώρα, όταν ε, υπολογίζουμε 200 ημέρες εργασίας, οι αποκεντρωμένοι φορείς υπολογίζουν 183 ημέρες εργασίας. Ε, υπάρχει μια διαφορά 14 ημερών. Ε, στη Γερμανία είναι κάτω από 10 ημέρες. Ο μέσος όρος ε, ημερών μπορεί κανείς να πουσιάζει Και στη Βαβαρία είναι 3,9% αυτό το ποσοστό. Ενδιέφερε να μου πείτε ε, πώς υπολογίζετε αυτά τα ποστά και πώς τα αξιολογείτε. Είναι πολλά κατά την άποψη είναι χαμένες μέρες εργασίας αυτές. Επίσης για την υπόθεση Τσίγκλερ είναι η ερώτηση παριθμών 34 που αφορά την υπόθεση Τσίγκλερ, η οποία πραγματικά είναι μια εντυπωσιακή ιστορία, όπου η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και ε, όσον αφορά την, επειδή υπήρξε μια συμφωνία όσον αφορά τις τιμές. Θα ήθελα να μας κάνετε μια πολιτική αξιολόγηση για την υπόθεση αυτή, μια πολιτική εκτίμηση, γιατί πραγματικά δεν είναι δυνατόν να, ισχύει κάτι να γίνεται κάτι τέτοιο. Όσον αφορά ε, την Όλαφ, ε, τις περιπτώσεις με τις οποίες ασχολήθηκε η Όλαφ, πόσες ήταν στην περίπτωση Τσίγκλερ. Και πραγματικά θα χαιρόμουν πάρα πολύ εάν μου λέτε ε, πότε ε, ε, να αναφερθεί στις κατεξουδότηση πράξη στο παράρτημα 10 για τις τρίτες χώρες. Γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα το οποίο έγινε στον, στον κανονισμό υπερσιακή κατάστασης. Και θα με διέφερε να μου πείτε τι γίνεται στην περίπτωση αυτή. Ευχαριστώ, πολύ. Ε, παρακαλώ τώρα να λάβουν ε, το λόγο οι εκπρόσωποι εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για την Άλντο Γιάν Μούλτερ. Ε, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομη η ερώτησή μου. Ξέρετε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές και θα ανανοηθεί βέβαια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν εσείς θα παραμείνετε, κύριε Σεύκοβιτς, πάντως, επί του παρόντος και γενικότερα αυτή την περίοδο έχουμε διάφορους εργαζόμενους στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι ψάχνουν να βρουν καλύτερες θέσεις εργασίας. Το ονομάζουμε αυτό παρασουτάζ στα γαλλικά. Είναι η διαδικασία του αλεξίπτωτου, όπου βασικά προσπαθεί ένας εργαζόμενος σε γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βρει μια καλύτερη, καλύτερα αμοιβόμενη θέση, να καταφέρει να προαχθεί κατά κάποιο τρόπο, ακόμα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να καταφέρει να εξασφαλίσει μια θέση προϊσταμένου μονάδος, διευθυντή, γενικού διευθυντή και το καθεξής. Ο Επίτροπος αναγνωρίζει την τάση αυτή και πώς θα μας διασφαλίσει τελικά ότι του χρόνου όταν για μία περίοδο δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος, δηλαδή από τον Ιούνιο στο Νοέμβριο 2014, μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι οι προαγωγές που θα γίνουν θα είναι πραγματικά δίκαιες και διαφανείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριο Μπάλστας έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να στηρίξω τα όσα είπε η συνάδελφος Γκρέσλε για τον κύριο Πετή. Νομίζω ότι πραγματικά υφίσταται μια ξεκάθαρη περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων, ακριβώς όπως είπε η κυρία Γκρέσλε. Και ως πρώην Γενικός Διευθυντής εργαζόμενος νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμίχθηκε στην περίπτωση Φίλιπ Μόρις και στη συνέχεια ανέλαβε μια πολύ σημαντική θέση στα πλαίσια μεγάλης κάπνο και τώρα τον βλέπουμε να εργάζεται στην ad hoc Επιτροπή Διοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Απάντηση λοιπόν επ' αυτού θα ήθελα και να απαντήσετε περισσότερο σε ερωτήσεις 44 ε, και τις ακόλουθες ε, όσον αφορά καταρχάς τα προϊόντα καπνού Ξέρετε ότι υπάρχει μια σύμβαση πλαίσιο όσον αφορά τον έλεγχο των προϊόντων καπνού και εκεί πέρα προβλέπεται τι, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα στο άρθρο 5 τους λομπίστες από τον κλάδο της καπνοβιομηχανίας, πώς μπορούμε να ελέγχουμε του ανθρώπου αυτού που ασκούν πίεση, γενικότερα τι ομάδε πίεση. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσετε λίγο πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση 43. Μα λέτε γενικά και αόριστα ότι έχουμε κάποιου κανόνε που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στον έλεγχο και την επιτήρηση των ομάδων επιρροή. Δεν νομίζω ότι γίνεται όμω κάτι τέτοιο τελό δημόσια και ανοιχτά και δεν έχω την εντύπωση ότι όλα καταγράφονται στο Μητρό Διαφάνεια. Επίση, η απάντηση που δόθηκε στην ερώτηση 44 είναι αρκετά αόριστη δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι επαφές που έχουν οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εκπροσώπους των ομάδων πίεσης και επιρροής. Αναφέρεστε εσείς σε κάποιες επαφές που είχατε, καθώς επίσης και με τον κύριο Βίλαρτ, αλλά αν καταλαβαίνω καλά, γίνεται λόγος για την ενδυνάμωση του λεγόμενου μητρώου διαφάνειας και θα έπρεπε ενδεχομένως το μητρό αυτό να γίνει υποχρεωτικό. Επομένως όλους οι σε ομάδες πίεσης να καταγράφονται, να καταχωρούνται σε αυτό το μητρό και να μπορούμε να παρακολουθούμε επακριβώς με ποιους έρχονται σε επαφή και τι ακριβώς κάνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ο έλεγχο αυτό, η διαφάνεια αυτή να υπάρχει όχι μόνο για τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά για όλο το προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έρχεται ενδεχομένω σε επαφή με εκπροσώπου ομάδων πίεση. Η σχετική ομάδα εργασία πότε θα ολοκληρώσει την εργασία τη. Αναφέρεστε γενικά στι επαφέ που είχατε με τον κύριο Βίλαντ. Θα θέλαμε ή δυνατόν να έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα πριν τι ευρωπαϊκέ εκλογέ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλα σχόλια από άλλε ομάδε. Ε, ποιος θέλει τώρα να μιλήσει, θέλετε εσείς, όχι. Ο, τότε δίνω το λόγο στον κύριο Επίτροπο. Να απαντήσετε παρακαλώ. Thank you uh, Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ε επανέρχομαι στο θέμα του κυρίου Μισελ Πετή. Έλαβα το μήνυμά σας, είναι σαφέστατο. Ε, ταυτόχρονα πρέπει να σας πω ότι το συζητάμε αυτό ακόμα σε εσωτερική διαδικασία εν ώψη ιδίως των ε, εξελίξεων του χρόνου. Ε, ποια θα είναι η σύνθεση της Επιτροπής Διοντολογίας, θα, θα αυξήσουμε τα μέλη, θα τα διατηρήσουμε ως έχουν και ποια θα είναι η καλύτερη σύνθεση ε, αυτής της Επιτροπής θέσατε το ερώτημα και μπορώ να απαντήσω εν μέρη για την επιλογή του Μισελ Πετή. Ήταν πρώην Γενικός Διευθυντής, ξέρει πώς εργάζεται η Κομισιόν, είχε, ε, ε, ε, έχερε του σεβασμού όλων και από την νομική, επιτροπή, η νομική υπηρεσία, έχει μια πολύ καλή νομική βάση και γνώσεις και σε όλες τις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή Δεοντολογίας υιοθετούσε μία απόφαση ή εξέδιδε μία ανακοίνωση εκείνος ως ε, νομικός εμπειρογνώμων ε, είχε ένα ρόλο να παίξει όμως ε, ας μην ξεχνάμε ότι η Επιτροπή Διοντολογίας έχει και άλλα καθήκοντα και η έγκριση, η υλοποίηση πολλών αποφάσεων γίνεται από κοινού με συναρμόδιους φορείς το, θέμα αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές. Ε, το συζητήσαμε και με τον διαμεσολαβητή και εξετάζουμε αυτή τη στιγμή πώς μπορούμε να δομήσουμε, να εδραιώσουμε ένα σύστημα όπου δεν θα υπάρχει καμία αμφισβήτηση ε, του ρόλου της Επιτροπής Δεοντολογίας. Επειδή του χρόνου θα έχουμε οπωσδήποτε, θα, θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ιδίως για την επιλογή και εξολόγηση των επιτρόπων. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα του κυρίου Στάες για τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και για συναντήσεις με το λόμπι του, του τομέα του καπνού. Πιστεύω ότι όπως είπατε, θα πρέπει οι συζητήσεις αυτές να γίνονται δημόσια, να ανακοινώνονται δημόσια, να τηρούνται πρακτικά που να είναι δημόσια προσβάσιμα και να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Σας διαβεβαιώ ότι όλα αυτά τα επενθυμίσαμε στο, στους υπαλλήλους μας και τα τονίσαμε αυτά στην ε, τελευταία εβδομάδα δεοντολογίας που έγινε πριν από δύο εβδομάδες. Είχαμε ένα σαφές διάγραμμα των κανονισμών για να αποφύγουμε συγκρούσεις συμφερόντων. Ειδικά όμως για αυτή την περίπτωση θα ε, έχουμε περαιτέρω κανόνες, επιπρόσθετους κανόνες από πλευράς του ΠΟΗ και πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Ε, γι' αυτό θα κάνω βεβαίως ό,τι μπορώ, θα σας διαβεβαιώ ότι αυτοί οι κανόνες θα γίνουν σεβασμοί, σεβαστοί. Ε, αύριο θα έχουμε στις 8.30 μία συνεδρίαση για τις προσλήψεις ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον Αντιπρόεδρο κύριο Βίλαν και άλλους συνεισηγητές αύριο στις 8.30 το πρωί. Πολλές φορές οι συζητήσεις μας είναι έντονες, θερμές, αλλά αυτό γίνεται επειδή θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι ακόμα καλύτερο, ακόμα ευρύτερο και ακόμα πιο διαφανές από ό,τι είναι τώρα πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα όπως έχει αποφασιστεί και να ολοκληρώσουμε το έργο της ομάδας υψηλών στελεχών πριν τελειώσει ο χρόνος. Διότι η βασική ιδέα είναι ότι τα συμπεράσματα των εργασιών αυτής της ομάδας θα υποβληθούν και στην ΑΦΚΟ και στην Ολομέλεια πριν σταματήσει τη εργασία του το Κοινοβούλιο πριν λήξει αυτή η θητεία. Άρα λοιπόν παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη αυτής της ε, έξεσης, το σχέδιο έκθεση. Είμαστε σε επαφή με τους συζητητέ και πιστεύω ότι θα το ολοκληρώσουμε όλα αυτά. Τρία άλλα θέματα τα οποία εγώ προσωπικά χειρίζομαι και έχω σχέση με τη διαφάνεια. Πρώτον είναι το μητρό διαφάνειας. Εκεί μαζί με τον Αντιπρόεδρο κύριο Βίλαν προσπαθούμε να φέρουμε με το μέρος μας και το Συμβουλίο. Μέχρι τώρα εκπρόσωποι του Συμβουλίου ε, λάβαναν μέρος ως ε, παρατηρητές στην ομάδα ψηλών στελεχών. Ε, θα συναντήσω την ερχόμενη εβδομάδα νομίζω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ σημαντικό το Συμβούλιο γίνει μέλος στην κοινή γραμματεία, συμμετέχει στην κοινή γραμματεία έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνεργασία σε αυτό το θέμα των θεσμικών οργάνων. Το, το έθεσα αυτό προς συζήτηση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και πιστεύω ότι θα προχωρήσει το θέμα ε, παρόλο που ορισμένα κράτη-μέλη έθεσαν ορισμένα ζητήματα νομικής φύσεως δύο άλλα προβλήματα τα οποία είναι σχετικά φρέσκα, καινούρια. Τουλάχιστον έχω πάρει πρόσφατες πληροφορίες. Ε, ε, έχει σχέση με τις νομικές ενώσεις στις Βρυξέλλες, διότι πολλές επικρίσεις ακούγονται επειδή καλυπτόμεσα από τους κανόνες διαφάνειας που καλύπτουν και τις επιχειρήσεις αλλά και τις συζητήσεις με νομικές πτυχές υπάρχει μία έλλειψη όσον αφορά τις εταιρείε νομικών, δικηγορικές εταιρείε νομικών εμπειρογνωμόνων. Ε, κάναμε λοιπόν μια πολύ ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων με τον, εκπρόσωπο, με τον εκπρόσωπο των νομικών δικηγορικών ενώσεων και ε, σας διαβεβαιώ ότι θα, θα αυξάνουμε συνέχεια την πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια. Για μένα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζουμε ότι συνεχώς μας επικρίνουν ότι αυτές οι δικηγορικές εταιρείες και το lobbying το οποίο κάνουν δεν καλύπτεται από το όλο πλαίσιο διαφάνειας, άρα πρέπει να βρούμε μια λύση. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι εδώ Υπησέρχονται και νομικά προβλήματα και συνταγματικά προβλήματα. Παραδείγματο χάρη Ισπανία υπάρχει συνταγματική υποχρέωση αποκάλυψης των πελατών των ε, εταιριών και ενώσεων αυτών. Ε, το τρίτο θέμα που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι, θα έλεγα, ε, η πρόσφατη παρουσία και στο μέλλον η παρουσία των Αμερικανικών νομικών εταιριών που θα έρθουν στις Βρυξέλλες. Έρχονται και εγκαθίστανται στις Βρυξέλλες με τα, μέσα στα πλαίσια της, ε, των διαπραγματεύσεων του TTIP. Uh, και ε, από τη στιγμή που καταχωρούνται αυτές οι εταιρείες ως δικηγορικές ή νομικές εταιρείες, ε, καταχωρούνται στην Ευρώπη, ε, στις Βρυξέλλες εδώ πρέπει πάλι να είμαστε προσεκτικοί και να ε, προσέξουμε αυτό το τομέα ε, στις Βρυξέλλες και ιδίως στο επιχειρηματικό τμήμα και να δούμε πώς ε, μπορούμε να αποφύγουμε επικρίσεις, διότι πολλές φορές ακούγονται πολύ αρνητικά σχόλια και μας λένε ότι δεν λειτουργεί καλά το πλαίσιο διαφάνειας διότι έχουμε δεν έχουμε αρκετό προσωπικό, έχουμε μόνο 37 υπαλλήλου και πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε αυτό το νέο φαινόμενο τη εγκατάσταση αυτών των εταιριών στι Βρυξέλλε των Αμερικανικών. Τώρα, αρχίζοντα αντίστροφα, θα απαντήσω πρώτα στον κύριο Μούλτερ όσον αφορά τους αλεξιπτωτιστές. Κύριε Μούλτερ, σας διαβεβαιώ ότι γνωρίζω πολλούς υπαλλήλου στα θεσμικά όργανα και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι Όσοι έχουν την καλύτερη κινητικότητα, έχουν δηλαδή εργαστεί σε διαφορετικά επίπεδα, σε διαφορετικές γενικές διευθύνσεις, μέσα στο, στο γραφείο επιτρόπων, εκτός γραφείων επιτρόπων. Είναι ακριβώς αυτά τα στελέχη που θεωρούνται ως οι καλύτεροι, ότι αποδίδουν βέλτιστα, είναι εξαιρετικοί υπάλληλοι, διότι έχουν καταφέρει να συλλέξουν όλη αυτή την εμπειρία εργαζόμενοι σε διαφορετικές υπηρεσίες, μονάδες, διευθύνσεις και με διαφορετικά ντοσιέ. Έχουν λοιπόν μία ευρεία ε, γνώση των θεμάτων και εμπειρία. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να θεωρούμε τα μέλη των γραφείων των επιτρόπων ε, ε, με κάποια, να, να τους κολλήσουμε μια αρνητική ετικέτα διότι πολλές φορές δεν μπορεί κανείς ποτέ να, να πάρει μια θέση στο γραφείο του επιτρόπου, ενός επιτρόπου αν δεν έχει ένα πολύ καλό ε, υπόβαθρο εργασίας και παρελθόν σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, ο, ο Επίτροπος ε, με, με, με ένα προσωπικό 30-40 ανθρώπων ε, μπορεί να ήταν αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης ή πρώην υπουργό ή υφυπουργός. Εγώ δεν έχω 40 ανθρωπων μπορει να ηταν αντιπροεδρος μιας κυβερνησης η πρωην υπουργος η υφυπουργος εγω δεν εχω 40 ανθρωπους στην υπηρεσία μου, έχω τρεις γραμματείς και άλλους 5-6 συνεργάτες. Λοιπόν, πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε ε, τις ε, δυνατότητες αυτών των ανθρώπων ανοιχτές και ε, καταλαβαίνω τη δική σας ανησυχία ότι πιστεύετε ότι άπαξ και λήξη θητεία του Κοινοβουλίου δεν θα σεβαστούμε τους κανόνες μας. Αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει διότι έχουμε ξεκάθαρους κανόνες για τις προαγωγές για τις καριέρες, την εξέλιξη μιας καριέρας μαζί με τη διεύθυνση προσωπικού θα ε, εξασφαλίσουμε την συμμόρφωση προς όλους τους κανονισμούς ε, και ε, θα εξετάσουμε προσωπικά κάθε προαγωγή, κάθε εξέλιξη καριέρας αλλά όπως σας είπα όσοι άνθρωποι εργάστηκαν ε, στο προσωπικό γραφείο ενός επιτρόπου ε, δεν πρέπει να έχουν μια αρνητική ετικέτα κολλημένη πάνω τους, διότι σας είπα ότι είναι αξιόλογα στελέχη. Ε, ορισμένες φορές στεναχωριέμαι που αυτομάτως υπάρχει κάποια αρνητική αντίδραση. Λέει, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια αντίληψη ότι άμα δουλεύεις για τον επίτροπο έχεις αμέσως ορισμένα προνόμια. Δεν είναι έτσι, αυτομάτως δηλαδή, είσαι προνομιούχος. Και ερχόμενη τώρα στην κυρία Γκρέσλε, θα επανέλθω πάλι στο θέμα της, το, των δαπανών μετακόμισης κλπ. Και... Ε, έχει αναφερθεί το θέμα αυτό σε διάφορες ε, περιπτώσεις και μετά από μακρές συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους συγητές ε, και, τις, και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την οποία πραγματικά αφορά πάρα πολύ αυτό το κόστος ε, είπαμε ότι αν θέλουμε να απλωστεύσουμε και να, τη διαδικασία και να εξοικονομήσουμε χρήματα θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον, μηχανισ, τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και να υπάρξει ένα όριο ούτω ώστε να μπορέσει να απλοποιηθεί τα πράγματα όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την εξοικονόμηση των χρημάτων και να υπάρχει δυνατότητα ενός πιο ξεκάθαρου ελέγχου του προπολογισμού για να είμαστε βέβαιοι ότι τα χρήματα αυτά δεν υπερβαίνουν το κατόφλιο αυτό. Και βεβαίως ε, η μελέτη θα ε, αυτή θα βασιστεί σε μια ε, καλή έρευνα της αγοράς. Τώρα όσον αφορά το επίδομα, την άδεια ασθενείας. Εδώ ε, έχω κάπως διαφορετικά στοιχεία, κάπως διαφορετικούς αριθμούς. Γιατί εάν δούμε τι γίνεται με αυτές τις αναρωτικές άδειε το 11 και το 12 οι απουσίες ήταν 3,8% και όταν ε, μιλάμε για απόλυτους αριθμούς εκφράζουν, αντιπροσωπεύουν 13 ημέρες αυτά τα ποσοστά. Ε, βεβαίως ε, μπορούμε να συζητήσουμε ε, για αυτά τα στατιστικά στοιχεία, αλλά εν πάση περιπτώσει αφορούν και τις Κυριακές. Είναι πρόκειται και σοβαρές περιπτώσεις ασθενείας. Εάν συγκρίνουμε τις, τα στοιχεία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε ότι στο Βέλγιο είναι περίπου 6%, στη Γερμανία είναι 4%. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λοιπόν κανένα πρόβλημα εάν ε, διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των ερωτικών αδειών, βεβαίως θα διενεργήσουμε τους ε, αντίστοιχους ελέγχους και θα διαπιστώσουμε κατά πόσο πράγματι υπάρχει ασθένεια ή ε, κατάχρηση, περίπτωση κατάχρησης. Τώρα, όσον αφορά τους απόλυτους αριθμούς και αναφέρομαι εδώ στα ποσοστά, θα αναφερθώ και εδώ, εδώ πάλι σε ποσοστά ε, σε σχέση με τους ελέγχους. Γιατί Καμιά φορά υπάρχουν αλλαγές ε, όσον αφορά τα νούμερα ε, των όσων απασχολούνται σε αυτές τις γενικές διευθύνσεις. Σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχουν αλλαγές στο οργανόγραμμα, στα οργανογράμματα τα οποία εγκρίνονται. Άρα λοιπόν ποικίλουν οι αριθμοί των απασχολούμενων ε, στις γενικές διευθύνσεις. Βεβαίως τώρα θέλουμε να υπάρξει μία μείωση του προσωπικού η οποία θα, βεβαίως θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στην Κομισιόν, γιατί όταν παρουσίασα για πρώτη φορά αυτή, αυτό το θέμα στη Γενική Διεύθυνση, του είπα ότι εάν θέλετε να προετοιμάσετε τη δική σας Γενική Διεύθυνση για την περικοπή προσωπικού, θα πρέπει να υπολογίσετε ένα 15%. Γιατί, γιατί το 5% φεύγει. Ε, είναι το 5% θα σας το πάρουμε γιατί θέλουμε να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία εντός της Κομισιόν ε, για το κατά πόσο χρειάζεται περισσότερα, μεγαλύτερο προσωπικό ή όχι. Και το 5% το θέλετε εσείς, το χρειάζεστε εσείς για να δείτε πώς θα τα καταναμίμετε τα χρήματα αυτά στην ίδια σας τη γενική, ε, ε, το ποστό αυτό συγγνώμη, στην ίδια τη γενική διεύθυνση. Άρα λοιπόν ε, είναι δύσκολο να εκφραστεί επακριβώς ο αριθμός αυτός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην περικοπή του προσωπικού για τους προϊστάμενους της κάθε μονάδας. Αλλά εάν ε, υπάρξει μεγάλη ζήτηση θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να σας θέσουμε στη διάθεσή σας αυτά τα στοιχεία. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε στα χέρια μας γιατί υπάρχουν διακυμάνσεις όπως σας είπα. Τώρα όσον αφορά τις συμβάσεις, ε, το έκτακτο, το, το προσωρινό προσωπικό, ο αριθμός αυτός ε, καλύπτει μόνο την επιτροπή. επιτροπή. Αυτός είναι ο μόνος αριθμός που έχω στη διάθεσή μου. Δεν νομίζω ότι οι εκτελεστικές υπηρεσίες καλύπτονται από αυτό το, αυτό το νούμερο. Και νομίζω ότι επίσης υπάρχει το θέμα το οποίο αφορά την περίπτωση, την υπόθεση Τσίγκλερ. Ξέρετε, είμαι σίγουρος, ότι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο υπάρχει τόσο ενδιαφέρον για αυτή την περίπτωση είναι το γεγονός ότι η εταιρεία Τσίγκλερ ε, τις επιβλήθηκαν πρόστιμα λόγω της συμπεριφοράς τους σε σχέση με, το νόμο περί, με τον κανονισμό περί καρτέλ. Ε, αυτή είναι απόφαση του δικαστηρίου. Ε, πληρώθηκε αυτό το πρόστιμο, άρα ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρξε μια παραβίαση. Και βεβαίως ε, υπήρξε και το αντεπιχείρημα εκ μέρους της εταιρείας, το οποίο έλεγε ότι το οποίο αναφερόταν στη συμπεριφορά των αξιωματούχων της Επιτροπής. Και το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε και πάλι από το δικαστήριο και στη συνέχεια ε, ε, έγινε, ασκήθηκε έφεση στην απόφαση. Νομίζω λοιπόν και ζητήθηκαν κάποιες αποζημιώσεις και νομίζω ότι για αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συζητιέται η περίπτωση αυτή μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τους αξιωματούχους της Επιτροπής, εμείς παραπέψαμε την υπόθεση αυτή στην Όλαφ και διεξήχθησαν κάποιες έρευνες. Σε τέσσερις περιπτώσεις ε, ασκήθηκαν ε, πειθαρχικά μέτρα, εφαρμόστηκαν πειθαρχικά μέτρα και ένα οδήθηκε σε περικοπή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Στη δεύτερη περίπτωση έγινε μια γραπτή μομφή και ε, στη τρίτη περίπτωση υπήρξε μια προειδοποίηση για μελλοντική κράτηση αυτών των αξιωματούχων. Άρα λοιπόν ε, πραγματικά αξιοποίησαμε όλες τις δυνατότητες που είχαμε στη διάθεσή μας και διεξήχθη πραγματικά λεπτομερής έρευνα και αυτό ήταν το αποτέλεσμα, η επιβολή αυτών των πειθαρχικών μέτρων. Κύριε Πίτροπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις λεπτομερείς αυτές απαντήσεις που μας δώσατε. Ένας ακόμα συνάδελφος θέλει να πάρει το λόγο, κύριος Μπραντμπορν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω από τι απαντήσει που έχετε δώσει μέχρι στιγμή όσον αφορά τι εκτελεστικέ υπηρεσίε, εκτελεστικού οργανισμού, θα ήθελα να αναφερθώ όλο ιδιαίτερω στι παρατηρήσει του κυρίου Στά, για τη σύγκρουση συμφερόντων. Στα πλαίσια του δικού σας χαρτοφυλακίου, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να γνωρίζω ποια μέτρα έχετε λάβει προκειμένου να μην υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων όσον αφορά τους διορισμούς που γίνονται σε εκτελεστικές υπηρεσίες. Θα θυμάστε ότι στο παρελθόν, όταν ασχοληθήκαμε με τα ζητήματα αυτά, είδαμε ότι υπήρχαν πολλές εικασίες για συγκρούσεις συμφερόντων και πολύ συχνά ακούμε τέτοιες κατηγορίες, τέτοιες εικασίες Γίνονται μάλιστα και άμεσα προς εμένα τέτοιες ε, κατηγορίες για τις ε, διαδικασίες πρόσληψης και διορισμού στις εκτελεστικές υπηρεσίες. Επομένως, στα πλαίσια των δικών σας αρμοδιοτήτων, ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν από εσά προκειμένου να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοιες συγκρούσεις συμφερόντων. Δεύτερον, Όσον αφορά πάλι τις εκτελεστικές υπηρεσίες, κάπου στο εγγραφό σας αναφέρεστε στο ότι ε, σε επίπεδο διευθυντικό το προσωπικό έχει παραμείνει σταθερό. Δεδομένου ότι έχουμε 37, δεν κάνω λάθος, τέτοιες εκτελεστικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να γνωρίζω αν έχετε περαιτέρω πληροφορίες να μας δώσετε για ενδεχόμενες περικοπές προσωπικού που έχουν γίνει στις υπηρεσίες αυτές και ενδεχόμενες μετακινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα κεντρικά γραφεία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις εκτελεστικές αυτές υπηρεσίες. Η κυρία Γκρέστα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπατε για αυτό το οικοδόμημα, Μισελ Πετή. Αναφερθήκατε στην ιδανική ε, σύνθεση τέτοια, αυτής της Επιτροπής. Ε, ας μην πούμε ιδανική, ας πούμε αξιόπιστη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αξιόπιστη η Επιτροπή αυτή, ε, διότι θα κατηγορηθεί για κακή διαχείριση. Εδώ και 1,5 χρόνο προσπαθούμε να παρακινήσουμε την Κομισιό να κάνει κάτι επιτέλους, διότι θέλουμε αξιόπιστες λύσεις. Δεν είναι ότι αυτό είναι το αγαπημένο μας θέμα και δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. Μας πυροβολούν οι απ' έξω, οι πολίτες και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να αριθμιστεί αυτό το συστήμα θέμα εφόσον ακόμα μπορούμε να το λύσουμε και να το ρυθμίσουμε. Γι' αυτό επισημούμε μια αξιόπιστη λύση. Τώρα αν είναι ιδανική μπορεί να πετύχει, μπορεί να μην πετύχει, αλλά το θέμα είναι να μην καθυστερούμε διότι... Ε, ακόμα ε, και στο, στον προηγούμενο προπολογισμό είχαμε συζητήσει το θέμα ε, της Επιτροπής Διαντολογίας και πώς συμπεριφέρεται σε περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων. Τώρα, πεκούνια και όλα. Ε, δεν έχω τίποτα προσωπικό κατά του ε, Μισελ Πετή, αλλά είναι θέμα ε, κακοδιαχείρισης. όλα αυτά νομίζω τα ο χειρισμός τους είναι πολύ προβληματικός. Εν συνεχή ερώτηση 43. Η Κομισιόν λέει ότι τα, το, εθνικό, ηθικό πλαίσιο της Κομισιόν συνάδει απολύτως με το, τους κανονισμού τη FCTC της ε, Σύμβασης Πλαίσιο για τον έλεγχο των προϊόντων καπνού από τον ΠΟΗ. Θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσετε ε, πού βασίζεται αυτή την απάντηση. Όσον αφορά επίσης ε, το προσωρινό προσωπικό, καλό θα ήταν να ξέρουμε και το μέσο όρο ε, των μισθών των προσωρινών αυτών υπαλλήλων. Εμένα ε, ε, μου υποβάλλονται πάρα πολλά παράπονα και θα ήθελα να ξέρω τα παράπονα είναι δικαιολογημένα. Ε, στο δημόσιο η πρόσληψη προσωρινών υπαλλήλων είναι πάντοτε προβληματική. Δεν θέλουμε να έχουμε να κάνουμε εδώ να αντιμετωπίζουμε χωριά ποτέμκιν από χαρτόνι δηλαδή τα οποία ντε και σόνι πρέπει να παραμένουν όρθια. Ε, ούτε είπα ότι το προσωπικό των, επιτρόπων έχει αρνητικές ετικέτες, αλλά ε, ε, μία, ένας διαγωνισμός ο οποίος κατά 80%, καλύπτει κατά 80% θέσεις και όχι το υπόλοιπο 20% μέσω διαγωνισμού, αυτό το βρίσκω πάρα πολύ προβληματικό και καθόλου δεν συμβάλλει στην αξιοπιστία μας. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η κυρία Παναγιώτοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, συγχαρώ τον Αντιπρόεδρο και ε, Επίτροπο κύριο Σεφτοβιτς για τις προσπάθειές του να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις αλλά και για την δέσμευση του έναντι του διαθεσμικού διαλόγου και των ε, ενδελεχών επαφών και συζητήσεων με τα εθνικά κοινοβούλια. Εγώ προέρχομαι από το κοινοβούλιο της χώρας μου και είχα την χαρά να συζητήσω με τον κύριο Επίτροπο τις διαθεσμικές σχέσεις με το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο μετά από την θέση ενισχύει της ε, συνθήκης. Είχαμε λοιπόν ε, τη χαρά να συζητήσουμε την ε, στρατηγική εστίαση στη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει λιγότερο ενδιαφέρον για την μετακίνηση υπαλλήλων που είναι ε, εμπειρογνώμονες και αν υπάρχει κάποια μείωση μετακινήσεων των υπαλλήλων αυτών προς τις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Ähm, ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Πίπερ και μετά ο κύριος Μούλντε. Έχω μια διευκρινιστική ερώτηση γιατί ο κύριος Μαγκορούτσα από το ελεγκτικό συνέδριο δεν πήρε ακόμα το λόγο. Ε, θα τον πάρει ή όχι. Ε, γιατί θα ήθελα να του οφείλω μια ερώτηση σε αυτόν ειδικά. Γιατί η απάντηση του Επιτρόπου ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είχα ερωτήσει πού προσλαμβάνουν οι Κομισιόν και το Ελεγκτικό Συνέδριο, από πού προσλαμβάνουν το προσωπικό τους. Και είπαν, είπε ως απάντηση ότι είναι στο πλαίσιο μια κοινή ε, εκπαίδευση την οποία κάνουν τα διαθεσμικά όργανα. Θα με ενδιέφερε πραγματικά να μας πείτε πόσο κοινή είναι αυτή η διαδικασία, πόσο αλληλένδετη είναι αυτή η διαδικασία. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω το ελεγκτικό συνέδριο πώς ε, προσλαμβάνετε εσείς το δικό σας ε, προσωπικό και αν υπάρχει μια κοινή εκπαίδευση για Κομισιόν και Ελεγκτικό Συνέδριο, κάποτε θα πρέπει να κληθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει επίσης μέρος, γιατί πραγματικά θα μπορούσαμε όλοι να αποτελέσουμε μια ευτυχισμένη οικογένεια, γιατί νομίζω ότι εγώ δεν είμαι επαρκώς καταρτισμένος. Ε, Μούλτερ. κατά από πόσο γνωρίζω ε, ε, ότι στο παρελθόν υπήρξαν ε, κάποιοι ισχυρισμοί ότι αν κάποιος εργαζόταν στο γραφείο ενός επιτρόπου, στο τέλος της θητείας δεν είχε πολλές πιθανότητες προαγωγής. Ε, ίσως αν η Επιτροπή μπορεί να μας παράσει κάποια στατιστικά στοιχεία θα ήθελα να τα δω. Εγώ δεν ε, ήθελα να, να μιλήσω αρνητικά για κάποια μέλη του πολιτικού γραφείου της Επιτροπής. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ε, δυστυχώς η ώρα έχει παρέλθει. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Επίτροπο και τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου να απαντήσουν τις ερωτήσεις. Και εγώ θα ήθελα να απευθύνω προς τον κύριο Επίτροπο και μια δική μου ερώτηση σε σχέση με τη σύγκρουση συμφερόντων. Ε, και ο ΣΑ εδώ έχει ε, εκπονήσει κάποια κριτήρια και ταυτόχρονα οι χώρες ε, μέλη παρακολουθούνται από αυτόν τον οργανισμό. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εδώ μέλος και παρόλο που όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του ΟΣΑ. Όσον αφορά το ζήτημα λοιπόν του, της εξωτερικής ε, παρακολούθησης της ε, Κομισιόν. Ε, συζητήθηκε μέχρι πρόσφατα το θέμα κατά πόσο η Κομισιόν δεν θα έπρεπε να γίνει η ίδια μέλος του ΕΣΑ. Δεν ξέρω, ίσως αν δεν μπορείτε να μου απαντήσετε τώρα θα ήμουν ευγνώμων για μια γραπτή απάντηση. Και ένα ερώτημα το έμεινε επίσης ανοιχτό ε, και ίσως ενδεχομένω θα μπορούσατε να το απαντήσετε και αυτό γραπτά, εάν δεν μπορεί να απαντηθεί εδώ προφορικά. Ποιο ερώτημα ήταν, ρωτάει ο κύριο Πρόεδρο η ερώτηση του κύριου Πίπαξ. Εάν δεν μπορείτε να την απαντήσετε, παρακαλώ, τώρα παρακαλώ να απαντηθεί γραπτά. Ωραία λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η τελευταία σας ερώτηση κύριε είναι σημαντική γιατί αναφέρεται ακριβώς στις εκτελεστικές υπηρεσίες. αλλά νομίζω ότι πρόκειται για υπηρεσίες που υλοποιούν το πρόγραμμα στις ε, Βρυξέλλες. Ε, κυρίως ε, πολιτιστικά ε, πολιτικές χορηγίες της Βρυξέλλες και αν υπάρχει εκεί μια σύγκρουση συμφερόντων, το πρόβλημα το οποίο γύρεται δεν είναι μεγάλο, γιατί το προσωπικό αυτών των υπηρεσιών ε, οφείλει να τηρεί τον κανονισμό. Αλλά νομίζω ότι εσείς ε, αναφερόσατε στους αποκεντρωμένους φορείς. Γιατί όταν μιλάμε για τους 33 οργανισμούς, αυτό το τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικός και ορθά είπατε ότι υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί και ε, ε, έχει ασκηθεί κριτική στην ε, έναντι της συμπεριφοράς των υπαλλήλων αυτών των αποκεντρωμένων οργανισμών. Αυτό έχει γίνει και έγινε ξεκάθαρο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συζήτηση σε σχέση με την αλλαγή του κανονισμού υπηρεσιακή κατάσταση. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι μια βελτίωση της διαχείρισης. Ε, και τι θέλουμε ακριβώ να γίνει σε σχέση με το ζήτημα τη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά του αποκεντρωμένου φορεί. Έχουν γίνει λοιπόν κάποιε διαβουλεύσει σε σχέση με το πώς θέλουμε να βελτιωθεί η διαχείριση και η πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων στους αποκεντρωμένους φορείς. Θα πρέπει να γίνεται ξεκάθαρα ούτως ώστε οι κανόνες αυτοί να ισχύουν για όλους, για το Διοικητικό Συμβούλιο, για τις Επιστημονικές ε, Επιτροπές και όλους όσους ε, μέχρι τώρα ε, δεν ήσαν υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες που ίσχυαν στο πλαίσιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Ε, για παράδειγμα, όσον αφορά την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και την αναγνώριση ενδεχόμενου κινδύνου, μελλοντικού κινδύνου ε, σύγκρουση συμφερόντων ε, και ποια, και θα έπρεπε να είναι τα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να λάβει κανείς. Αλλά εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω ότι αυτοί οι αποκεντρωμένοι φορείς δεν διευθύνονται από την ε, Κομισιόν, αλλά από τα διοικητικά του συμβούλια. Και ε, βεβαίως κατανοώ το ότι μου απευθύνεται αυτές τις ερωτήσεις που δικαιολογούνται, νομοποιούνται πολιτικά, αλλά ε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, για παράδειγμα, σχετικά αφορά τη συγχώνευση αυτών των οργανισμών της Europol με κάποιον άλλο φορέα. Ε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, γιατί είναι τα διοικητικά συμβούλια αυτά τα οποία αποφασίζουν. Εμείς μπορούμε να υποβάλουμε βεβαίως κάποιο, μια ξεκάθαρη δέσμη κανόνων οι οποίοι εφόσον τηρούνται θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της πρόληψης μελλοντικών συγκρούσεων συμφερόντων. Και βεβαίως ε, είμαι στη διάθεσή σας για μια σχετική συζήτηση αυτών των κανόνων, εάν θέλετε και πριν από τα Χριστούγεννα μπορώ να σας αποστείλω για να στήσουμε τον Ιανουάριο. Τώρα, όσον αφορά τη συνεργασία με τον ΩΣΑ, ε, πραγματικά είναι μια πολύ σωστή και χρήσιμη ιδέα. Ε, και εγώ ίδιος ε, συμμετείχα σε μια τέτοια συζήτηση στο Παρίσι, όπου η δική μας πρακτική αξιολογήθηκε θετικά και ζητήθηκε η δική μας γνώμη για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια, για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων και πώς μπορούμε να αντλήσουμε δάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές ε, μιας από τις καλύτερα λειτουργούς οικονομίες του κόσμου. Ε, όλες οι χώρες μέλη είναι του, όλες οι χώρες μέλη της Ένωσης είναι μέλη του ΟΣΑ και ε, είναι γνωστό ότι ασκούνται τέτοιες ε, πιέσεις για προσχώρηση στον ΩΣΑ. Είναι γνωστές επίση οι διπλωματικές δυσκολίε από την άλλη. Άρα λοιπόν ε, είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανείς τις ε, πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά βεβαίως η, η όφηση, η ανάγκη για αύξηση διαφάνειας υφίσταται και θα υπάρξει μια σχετική πρόσκληση από την ομάδα που εργάζεται για την βελτίωση της διαφάνειας. Ο κύριος Μάλτερ είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή αντιμετώπιση των μελών του γραφείου, των γραφείων των επιτρόπων. Εγώ θα έλεγα ότι πάλι υπάλληλοι ότι πάλι αυτοί χαίρουν ε, μεγάλης γιατί συγκεντρώνουν πολύτιμες εμπειρίες, γιατί βεβαίως συνεργάζονται σωστά, ε, στενά με το πολιτικό κομμάτι της, ε, στο πλαίσιο από τη, διαδικασία διαδικασίας αποφάσεων της Κομισιόν. και βεβαίως ε, δεν θέλουμε να υπάρξει μια ε, κατάχρηση ε, της εξουσίας τους. Of, uh, on... Να περάσω τώρα στην ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε όσον αφορά τα προϊόντα καπνού. όσον αφορά την καπνοβιομηχανία και τις επαφές που έχουμε μαζί τους. Όπως σας είπα και πριν από λίγο, ένας από τους κανόνες μας εξηγεί το πώς θα πρέπει εμείς να συμπεριφερόμαστε όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους εκπροσώπους της καπνοβιομηχανίας. Πρέπει προφανώς να τηρούμε τους κανόνες αυτούς πρέπει να ευαισθητοποιούμε όλους τους υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με τις επαφές αυτές. Και αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Αν συμβεί κάτι το οποίο ξεφεύγει από τους κανόνες αυτούς, αν θεωρείτε εσείς ότι δεν έχουμε τηρήσει κατά κάποιο τρόπο τα κριτήρια αυτά και αν εμπλέκεται τελικά στην παρατυπία αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προφανώς θα πρέπει να λάβουμε δράση προκειμένου να τηρούνται εκ νέου οι κανόνες αυτοί και να υπάρχει μια γενική συμμόρφωση με αυτούς. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Παναγιώτοβα, με συγχωρείτε, συνεχίζει ο επίτροπο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ θετικά σας λόγια, καθώς επίσης και για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε όταν ήσασταν επικεφαλής της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλγαρίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πάρα πολύ καλή επαφή και με τα κράτη-μέλη αυτά καθ' αυτά. Το βλέπουμε και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις τις διαδικασίες επί παραβάση. Μπορούμε να αποφεύγουμε τις διαδικασίες αυτές να κερδίσουμε πολύ πολύτιμο χρόνο. Πιστεύω λοιπόν ότι κατά διάρκεια ιδίω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να έχουμε πολύ θετικέ επαφέ με τα κράτη-μέλη και με κάθε κυβέρνηση όσον αφορά το ζήτημα τη οικονομική διακυβέρνηση. Σε ορισμένε βέβαια περιπτώσει, ο συντελεστής διόρθωσης είναι ο καθοριστικός τελικά παράγοντας που ε, μας καθιστά εμάς ε, λιγότερο ελκυστικούς αν θέλετε. Στη Σλοβακία ο στελεστής αυτός, αυτός είναι 8%, στη Βουλγαρία χαμηλότερος ενδεχομένως. Επομένως, αν ε, βρίσκεται κανείς στις Βρυξέλλες και εργάζεται στις Βρυξέλλες και του προταθεί να πάει να εργαστεί στη Βουλγαρία με μια μείωση της τάξης του 20%. Καταλαβαίνω βέβαια ότι η κατάσταση αυτή δεν θα είναι ιδιαίτερα ελκυστική δεν μπορώ όμω εγώ να κάνω κάτι γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει εγκριθεί ω κανόνα στα πλαίσια του κανονισμού υπηρεσιακή κατάσταση και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε δίκαιες αποδοχές για όλους τους εργαζομένους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε βρίσκονται στις ε, Βρυξέλλες, είτε βρίσκονται σε άλλες πόλεις της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τηρούμε ουσιαστικά το στελεστή αγοραστικής δύναμης και βάσει αφού του στελεστή προσαρμόζουμε τις αποδοχές. Πρόεδρος. Δύο συνάδελφοι θέλουν να πάρουν εκ νέου το λόγο. Ερώτηση θέλετε να υποβάλλετε προς τον Επίτροπο ή προς τον εκπρόσωπο του Λεπτικού Συνεδρίου. Προς τον Επίτροπο, παρακαλώ. Πρώτα η κυρία Γιάλα Σέντερ και συνέχεια ο κύριος Μούλτερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με την παρέμβαση του Επιτρόπου κύριου Σεύκοβιτς, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε απέναντι σε μια εκθέση του λεκτικού συνεδρίου και θα πρέπει να τους συγχαρούμε γιατί πραγματικά τριπλασίασαν τις, τον έλεγχο των συναλλαγών σε σχέση με το, την, την προηγούμενη χρονιά και πέτυχαν αυτό το 0%. Άρα θα πρέπει να τους συγχαρούμε. Ωστόσο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σε σχέση με τις εκτελεστικές υπηρεσίες θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Επίτροπο γιατί δεν νομίζω ότι όλοι έχουμε την ίδια γνώμη. Εάν η Επιτροπή είχε επαρκή χρηματοδότηση για να ε, προσλάβει βάση συμβάσεις αόριστης διάρκειας ε, τους υπαλλήλους των εκτελεστικών υπηρεσιών θα προσλάμβανε έκτακτους ε, προσωρινούς εργαζόμενους. Δεύτερον, σε σχέση με την ε, δεοντολογικό κώδικα, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σεφκοβίτς κατά πόσο... Ε, το εξής, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε έναν γενικό πλαίσιο δεοντολογίας. Να μην υπάρχει αυτή η κατάτμιση, αλλά να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για όλους τους ε, εργαζόμενους εν σχέση με τα ενδεχόμενα προβλήματα σύγκρουσης συμφερόντων και με τον, ε, σχέση με τον ΩΣΑ. Νομίζω θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα αυτή να έχουμε ένα ε, γενικό πλαίσιο δεοντολογικού κώδικα που θα κάλυπτε όλες τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ κύριε Μούλτερ. Κύριε Μούλτερ. Yeah. please, κάπως που ο Επίτροπος ερμήνευσε διαφορετικά την ερώτησή μου. Εγώ δεν ζήτησα μία δίκαιη μεταχείριση του προσωπικού του, των γραφείων των επιτρόπων. Εγώ ζήτησα μία θεμητή και δίκαιη κρίση και αξιολόγηση όλων, όλου του προσωπικού, όλων των υπαλλήλων. Μάλιστα, ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Δίνω το λόγο πάλι στον κύριο Επίτροπο και μετά στον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όταν μιλάμε για τη σύγκρουση συμφερόντων, όπως σας είπα ήδη, θα έχουμε αρκετές συζητήσεις επ' αυτού του χρόνου. Αλλά είναι σαφές ότι θέλουμε να βελτιώσουμε ορισμένες διαδικασίες στην Κομισιόν. Και αυτό τα, αυτές οι βελτιώσεις πρέπει ήδη να ληφθούν υπόψη από τις υπηρεσίε και τους φορείς. Θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη δήλωση ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων όταν εισέρχεται κανείς στην υπηρεσία και θα πρέπει να υπάρχει μια απογεγραμμένη δήλωση όταν κανείς φεύγει από την υπηρεσία και εισέρχεται στην συνταξιοδοτική περίοδο. Πρέπει κανείς να είναι σαφέστατος και ειλικρινής όσον αφορά τη συμπεριφορά, ε, την ε, μελλοντική εργασία, την οποία θα επιτελέσει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις έναντι των ε, θεσμικών οργάνων σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται ε, να υπάρξει ε, μια σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να αποτανθεί κανείς στην Κομισιόν και να ζητήσει μια γνωμοδότηση και βάσει αυτού η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να ε, μην εγκρίνει την υποψηφιότητα και να απορρίψει τον υποψήφιο. Πιστεύω ότι αυτή η γραμμή είναι σαφής, θα ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα τα οποία σας ε, στοχεύουν στη βελτίωση, δεν μπορώ να σας τα αναφέρω όλα, αλλά έχουμε υπόψη μας να δημιουργήσουμε ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου που θα ωφελήσει την απόδοση όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Σχετικά με την ερώτηση για τις έκτακτες ή προσωρινές προσλήψεις είναι πολύ δύσκολο να σας δώσω μία ε, οριστική απάντηση για το ποια, είναι, ποια φύση της εργασίας είναι καλύτερη. Ε, εξαρτάται. Ορισμένοι άνθρωποι προσλαμβάνονται βάσει ε, ε, δικαίου, βάσει συμβασιακού δικαίου του Βελγίου. Άλλοι χρειάζονται εκτάκτος, άλλοι χρειάζονται προσωρινά για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Άλλες φορές αντικαθιστούν κάποιον άλλον υπάλληλο, ιδίως σε υποστηρικτικές υπηρεσίες όπου Χρειάζεται απλώς μία αντικατάσταση ενός υπαλλήλου για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, θα δώσω λοιπόν μία, ε, το να δώσω μία και μόνο απάντηση σε όλες αυτές τις νομομένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά εμείς ε, θέλουμε να κριθούμε ως καλοί εργοδότης και ξέρω ότι και εμείς και το Κοινοβούλιο πάντοτε εξετάζει ε, τη δυνατότητα να προσφερθεί μια σωστή, σταθερή θέση εργασίας που να υπόκειται σε όλους τους κανόνες ε, ενός υγιεινού και σωστού εργασιακού περιβάλλοντος. Κύριε Μούλτερ, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη ε, αν παρερμήνευσα τα σχόλιά σας. Σημείωσα το, τη θέση σας και βεβαίως ε, θέλουμε και εμείς όλοι οι υπάλληλοι να κρίνονται ισότιμα και δίκαια. Και αυτή είναι η θέση μας. Σας ευχαριστώ που τονίσατε αυτό το ζήτημα και θα το σημειώσω και για προσυζήτηση ε, στην έδρα μου, στην Κομισιόν. Ο Πρόεδρος. Τώρα δίνω το λόγο στα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να σας εξηγήσω ορισμένα πράγματα και να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Σαπίπερ, ο εισηγητής, για το πώς έχει το σύστημα πρόσληψη στο λεκτικό συνέδριο. Όπως και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, συμμεριζόμαστε και μοιραζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υπηρεσία έψο, την υπηρεσία επιλογής κοινοτικού προσωπικού μέλη του ελεκτικού συνεδρίου συμμετέχουν ως κριτές, ως εξεταστές στην έψο και κατά αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν και με την εμπειρία που έχουν στον τομέα του ελέγχου. Περνάμε στη συνέχεια στο στάδιο της πρόσληψης, η οποία όμως δεν γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την έψο αυτή καθ' αυτή, αλλά από το ίδιο το ελεκτικό συνέδριο βάσει του κανονισμού μας. Καλούμε δηλαδή τους υποψηφίους για συνέντευξη, συστήνεται μια εξταστική επιτροπή, μια κριτική επιτροπή, αξιολογεί το κάθε υποψήφιος ξεχωριστά και στη συνέχεια αποφαίνεται το ελεκτικό συνέδριο για το ποιος τελικά θα επιλεγεί και είναι υπεύθυνο στη συνέχεια το ελεκτικό συνέδριο για τη μετέπειτα εξέλιξη της σταδιοδρομίας του νεοπροσληφθέντα. Να σας πω ακόμα ότι μολονότι δεν έχω στα χέρια μου συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα, το προσωπικό του ελεγκτικού συνεδρίου πρέπει προφανώς να έχει μια σημαντική πρώτερη εμπειρία στον τομέα πολλοί προέρχονται από την ιδιωτικό τομέα, από ελεγκτικές δηλαδή εταιρείε ή από άλλες εταιρείε που έχουν ε, χρηματοπιστωτικά ελεγκτικά καθήκοντα. Πολλά πάντως μέλη του προσωπικού μας προέρχονται και από ανώτατα δικαστήρια ή τα ίδια τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια των κρατών μελών. Άλλοι πάλι προέρχονται από το δημόσιο κλάδο, το δημόσιο τομέα των εθνικών των κρατών μελών, με συγχωρείτε. Το σύστημα πρόσληψης πάντως και επιλογής είναι διαφορετικό από το σύστημα εκπαίδευσης και περαιτέρω κατάρτισης των εργαζομένων μας. Ελπίζω να διευκρινίσει και κατά αυτόν τον τρόπο το ζήτημα το οποίο έθιξε ο κύριος Πίπερ. Ευχαριστούμε πολύ. Για να συνοψίσουμε τώρα λόγο, για να συνοψίσουμε τώρα δίνουμε το λόγο στον εισηγητή εφόσον επιθυμεί να πάρει το λόγο. Κύριο Πίπερ. Ναι, ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά μια πολύ καλή απάντηση. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται, υπόθηκε τελικά ότι είναι μια κοινή διαδικασία και θα μα ενδιαφέρει να μου αναφέρετε συγκεκριμένα τα ποσοστά. Αλλά θα πρέπει αυτό να το διευκρινίσουμε με το ελεγκτικό συνέδριο. Λοιπόν, τέθηκαν μια, τέθηκε μια μια σειρά από ερωτήματα και βεβαίως ε, κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις ε, έμειναν ανοιχτές. Θα υπάρξει λοιπόν ένας δεύτερος ε, κατάλογος εκείνων των ερωτήσεων οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί και πρόκειται να το συζητήσω σχετικά με τους συντονιστές. Ευχαριστούμε πολύ και εδώ ε, θα ανούμε στο τέλος αυτής της συζήτησης με τον Επίτροπο κύριο Σεύκοβιτς. Κύριε Σεύκοβιτς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ακριβείς σας ε, απαντήσεις στο μέτρο του δυνατού βεβαίως. Και ε, αυτή ήταν η πρώτη σας επίσκεψη εδώ σε αυτή την Επιτροπή και θα ήθελα να επαναλάβω το, το είπα στην εισαγωγική μου παρουσίαση. Σας συγχαίρομαι πραγματικά για το 0% ποσοστό σφαλμάτων. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί. Πραγματικά θερμά συγχαρητήρια γι' αυτό. Thank you.